Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, επαναλαμβάνουμε τη συνεδρίασή μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας δείξω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι παρόν σήμερα το πρωί. Θα χρειαστεί από τις 4.30 να ξαναλείψω για να συμμετάσχω στην ε, συνεδρίαση των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων που θα συζητήσει τις ε, πολιτείς ε, δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ τον George Lyon και για τις συνεδρίες των συντονιστών τη Utah Hawk που ανέλαβαν τα καθήκοντα προεδρίας. Ε, θέλω να χαιρετήσω τον Γιάν Μιούλτερ και μία ομάδα επισκεπτών από το Πανεπιστήμιο του Βάρνινγκ που έχει προσκαλέσει ο Γιάννη που είναι ο πιο διακεκριμένος φοιτητή ε, του Πανεπιστημίου αυτού, οπότε τους καλωσορίζουμε. Είναι πολύ ε, ενθαρρυντικό για μας που ενδιαφέρονται οι πολίτες της Ευρώπης τόσο πολύ ώστε να έρθουν εδώ στην έδρα μας, στις Βρυξέλλες. Όπως θα σας είπε ο Γιάνν, ότι αν δεν μπορείτε να έρθετε και αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε σπίτι σας, μπορείτε να ε, παρακολουθήσετε από την ε, τηλεόρασή σας ή από τον υπολογιστή σας τη συνεδριά της Επιτροπή Προπολογισμών που είναι πάντα συναρπαστικέ. Θα έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Έχετε παρατηρήσει, όχι. Ε, οι ψηφοφορίες θα αρχίσουν στις 4.30. Οπότε σας παρακαλώ στις 3.30 να είστε παρόντες με τις κάρτες σας για να μπορέσουν να γίνουν οι ψηφοφορίες σήμερα. Έχετε στα νέα ε, της Επιτροπής Αλέχου του Προπολογισμού της ανακοινώσεις του Προέδρου. Κατά τη συνεδρία στις 12 Μαρτίου οι συντονιστές αποφάσισαν να ορίσουν τον συνάδελφο Ντέρεκ Βόγγεν εισηγητή για τη γνωμοδότηση επί της εκθέσεως για τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών περιορισμών για ε, των, των δημοσιονομικών περιορισμών επί της ε, απορρόφησης των διαρθρωτικών πόρων. Ο κύριος Βόγγελ, που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας, ε, θα είναι και ο συντάκτης αυτής της γνωμοδότησης. Όσον αφορά την αποστολή αντιπροσωπείας στην Σερβία και το Μαυροβούνιο, τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέλεξαν τον Σαλβαδόρ Γαρίγα επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Συγχαίρουμε τον Σαλβαδόρ. ο οποίος περιμένει να το συγχαρούμε λοιπόν για να μπει στην αίθουσα γιατί είναι ιδιαίτερα μετριόφρον. Σήμερα το πρωί ασχοληθήκατε με τη δημόσια ακρόαση για τη χρηματοδότηση της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Να περάσουμε λοιπόν τώρα προτείνω στο σημείο 7 που είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2014. Η εισηγήτρια είναι η Αν Γένσεν Θέλετε να μας πείτε τι έγινε χθες στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνεδριάσαμε για πρώτη φορά. Ήσασταν και εσείς παρόν για τον προπολογισμό του 2014. Πρώτη συνάντηση λοιπόν των τριών θεσμικών οργάνων. Με βάση τις καθευτήριες γραμμές λοιπόν ε, συζητήσαμε που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο τη βδομάδα που μας πέρασε. Όπως θα θυμάστε, αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές τόνιζαν ότι καλούμε την Επιτροπή να μας κάνει προτάσεις που να ανταποκρίνεται στις προτάσεις της ίδιας της Κομισιόν για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την νομική βάση όσο δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των τριών οργάνων επί των πολιετών προοπτικών. Επιπλέον, οι καθευτήριες γραμμές ε, ασχολούνται και με τις πληρωμές που δεν θα θέλαμε να αναλάβουν και τους απλήρωτους λογαριασμούς του 2013 και του 2012. Ακόμη και αν υπάρξει ένα big bang διορθωτικού προϋπολογισμού που να φτάνει μέχρι το όριο του 2013. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη και αν υπάρξει τέτοιος προϋπολογισμός, θα υπάρξει μάλλον ε, έλλειμμα, γιατί δεν έχουν προβλεφθεί επαρκή ποσά για τις πληρωμές. Το αναφέραμε λοιπόν αυτό στην Επιτροπή και το Συμβούλιο και επιπλέον τονίσαμε ότι το κεφάλαιο 4 του προπολογισμού του 2014 θα πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων, τις πολιτικές μας δηλαδή προτεραιότητες. Νομίζω ότι Υπάρχει μια κοινή βάση μεταξύ των ε, τριών θεσμικών οργάνων, αλλά βέβαια παίζουν ρόλο και λεπτομέρειες. Ξέρω ότι και ο κύριος Λαβία έχει την άποψή του επ' αυτού, αλλά κατά τη δική μου ε, υπάρχει ασάφεια στην άποψη της Κομισιόν για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Δεν θα επιληθεί συντόμω το θέμα αυτό. Ρωτήσαμε επίσης ε, σε ποια βάση βασίστηκε η Επιτροπή για να κάνει αυτές τις προτάσεις. Δεν πήραμε σαφή απάντηση, αλλά μας είπαν ότι θα υποβάλουν τις προτάσεις τους επί του προϋπολογισμού ή στις 16 ή στις 30 Μαΐου. Ίσως λοιπόν τέλη Μαΐου, που είναι και η πιο πιθανή ημερομηνία, να έχουμε μια ιδέα. Θα αργήσουμε λοιπόν. Η Ιρλανδική Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε, εξέφρασε την ε, βούλησή της να συζητήσει το θέμα αυτό, να προσπαθήσει να βοηθήσει στην εξέβρεση λύσης αλλά είναι σαφές ότι επίσης εμένει στη γραμμή του Συμβουλίου. Στη γραμμή αυτού που αποκαλούν ε, λογικό προϋπολογισμό. Ε, χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις ε, αλλά έχουν διαφορετική έννοια. Όταν μιλάνε για παράδειγμα για τους διάφορους οργανισμούς, όλοι λέμε ότι πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους, αλλά όχι πάνω από ό,τι μπορούν να δαπανίσουν. Και εμεί συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πόροι για τους οργανισμούς. Αλλά για μια σειρά ε, οργανισμούς βλέπουμε ε, περίεργες περικοπές του Συμβουλίου. Για παράδειγμα, ε, οι οργανισμοί επιτήρηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα να υφίστανται περικοπές στην παρούσα συγκυρία. Τέλος πάντων. Πολύ καλά πήγε, πολύ καλή συζήτηση, αλλά υπάρχουν σοβαρές διαφορές ερμηνείας και σοβαρή έλλειψη ε, σαφήνειας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ αν όπως είπε και η Αν, λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εκτέλεσης του 2013 και των πιστώσεων πληρωμών. Ο Τζοβάνι, ο εισηγητής μας για το 2013. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εχθές Στη διάρκεια του τρεμερούς διαλόγου φυσικά έγινε λόγος για τις πληρωμές του 2013 και προφανώς ε, εξετάστηκε το θέμα των διορθωτικών προπολογισμών. Ο πρώτος διορθωτικός προϋπολογισμός έχει όντως ήδη προταθεί από την Κομισιόν που τον ανέκρινε το σύνολο των επιτρόπων στις 18 πριν από δύο μέρες δηλαδή και αφορά την ε, ένταξη της Κροατίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη της Κροατίας το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Επ' αυτού προφανώς το Συμβούλιο θα ξεκινήσει τον ε, προβληματισμό του και φυσικά θα πρέπει να πάρει θέση και το Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι από τη δική μας άποψη εφόσον ε, δεσμεύεται από πρόβλεψη της συνθήκης σε σχέση με τον ε, διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 1, η μόνη δυνατότητα είναι από πλευρά των κρατών μελών να δοθούν ε, φρέσκοι επιπρόσθετοι πόροι για να καλυφθεί ο διευθυντικό προπολογισμό αυτό. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η συζήτηση στο Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το στοιχείο και στη συνέχεια θα ενεργήσουμε. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να μειώσει όσο γίνεται το χρόνο εξέτασης ε, αυτού του διευθυντικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η προσχώρηση της ε, Κροατίας προβλέπεται για την 1η Ιουλίου και πρέπει εγκαίρως να προβλέψουμε το κλείσιμο της διαδικασίας. Η άλλη πτυχή αφορά τις πληρωμές του 2013. Όλοι γνωρίζετε την κατάσταση. Συνδέεται με το γεγονός ότι πέρυσι για να κλείσει ο προϋπολογισμός μια μεγάλη εφευρετικότητα, ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι εντόπισε μια νέα κατηγορία προϋπολογισμού, δηλαδή της ε, ε, εκρεμής ε, ανάγκης που μέσα στην οικονομική κουλτούρα προϋπολογισμού της Ευρώπης δεν είχε μπει ως όρος στην στο, στο λεξικό, αλλά φυσικά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη την αυτή κατηγορία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτή που είναι η κοινή δήλωση υψηλού επίπεδου που έγινε πέρσι ανάμεσα στις, στα τρία θεσμικά όργανα, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες πληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους. Είναι σαφές λοιπόν ότι χρειάζεται, όπως και στην ε, δήλωση αυτό προβλέπεται, ε, χρειάζεται λοιπόν ένας διορθωτικός προπολογισμός από την αρχή του έτους που θα λάβει υπόψη τις ανάγκες. Και από αυτού η Κομισιόν μας είπε ότι ΣΥ και ότι θα εγκρίνει η πρόταση πιθανότατα στις 27 Μαρτίου και είναι το περίφημο Big Bang στο οποίο αναφέρθηκε η συνάδελφος Γένσεν. Το περιμένουμε και ευχόμαστε ως Κοινοβούλιο η πρόταση διευθυντικού προϋπολογισμού να είναι συνεπής σε σχέση με τις απαιτήσεις πληρωμών του έτους που υπό το φως των εκτιμήσεων που έγιναν ε, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κομισιόν θα μπορέσει να το επανεξετάσει όσο γίνεται πιο σύντομα για να έχουμε πιο συγκεκριμένες ενδείξεις και μας λένε λοιπόν ότι προφανώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη ε, πιστώσεων πληρωμών. Ήδη από πέρσι οι εκρεμείς ε, ανάγκες, δηλαδή λογαριασμοί που έφτασαν στις 31 12 του 12 ε, βλέπουμε ότι λείπουν 16,2 δις ευρώ που μένουν ακάλυπτα. Περιμένουμε λοιπόν σαφώς από την Κομισιόν έναν διορθωτικό προϋπολογισμό συνεπή με τις απαιτήσει συνέχισης των προγραμμάτων, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ξαναδούμε ποια είναι η ομαλή διεξαγωγή και η υλοποίηση των προγραμμάτων και να επανεξετάσουμε τις δεσμεύσεις μας ώστε να μειώσουμε τις δαπάνες. Αυτό όμως δεν το ευχόμαστε ως Κοινοβούλιο. Εμείς θα θέλαμε όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί να μπορέσουν να συνεχιστούν όπως ξεκίνησαν να μπορέσουν να συνεχιστούν. Αλλά για να γίνει αυτό διαπιστώνουμε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη επιστώσεων πληρωμών. Και γι' αυτό Ευχόμαστε το τόσο αναμενόμενο Big Bang και που η Κομισιόν θα μας παρουσιάσει μετά από τις 27 να είναι στο, στάσος, στο ύψος των ε, απαιτήσεων για τις πληρωμές. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πιστεύω λοιπόν οι δύο εισηγητέ μας παρουσίασαν πολύ καλά την κατάσταση. Αυτός ο τριμερής διάλογος, όπως είπαν, ήταν η ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων και για επαλήθευση του πνεύματος υπό το οποίο εργάζονται οι εταίροι μας. Για να δούμε το πρόβλημα από χρονολογική ε, άποψη, να δούμε όσον αφορά τις συνέπειες ε, της δημοσιονομικής της ένταξης της Κροατίας που προβλέπεται για την 1η Ιουλίου και ταυτόχρονα για τεχνικούς λόγους αλλά κυρίως για πολιτικούς λόγους είναι ο καλύτερος τρόπος για να ευχηθούμε το καλωσόρισε στο νέο μας εταίρο. Θα θέλαμε ιδιαίτερα από πλευράς του Κοινοβούλου, το επιθυμούμε και το είπαμε, να έχουν ε, γίνει όλες οι απαραίτητες δημοσιονομικές προβλέψεις που θα επιτρέψουν στην Κροατία να εφαρμόσει όλες τις κοινωτικές πολιτικές από την 1η ε, Ιουλίου 2013. Για την ώρα το Συμβούλιο δεν έχει εξετάσει την πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού υπαρθμών 1 που είναι αφιερωμένο στην Κροατία και που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω την εντύπωση ότι τα νούμερα που προτείνει η Κομισιόν θα αμφισβητηθούν. Φυσικά, εμείς επιμείναμε από πλευράς μας ώστε τα ανώτατα όρια να προσαρμοστούν τουλάχιστον όσον αφορά τις λειτουργικές πιστώσεις. Ε, για τις διοικητικές επιπτώσεις θα το, πρέπει να το δούμε, αλλά να υπάρξει μια προσαρμογή των ανώτατων ορίων είναι πρόταση της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και σε λίγο θα γνωρίζουμε επί ποιας βάσης ε, βρίσκεται το Συμβούλιο. Όπως είπε ο εισηγητής μας, ε, εμείς επιμείναμε ώστε το Συμβούλιο να μην ε, χάνει χρόνο. Θα έλεγα να μην ε, καθυστερήσει, να μην χρονοτριβήσει, ιδιαίτερα με βάση αυτόν τον κανόνα των 8 εβδομάδων, για να μπορέσουν τα εθνικά κοινοβούλια ενδεχομένως ε, να δείξουν την αρχή της επικουρικότητας. Αυτή δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση και πιστεύω πως θα μπορέσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να αποφασίσει σύντομα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει το Κοινοβούλιο μας να είναι σε θέση να κάνει τελική ψηφοφορία όσον αφορά το διευθυντικό προπολογισμό το αργότερο τον Ιούνιο. Όσον αφορά τις πληρωνές του 2013, την εκτέλεση του προπολογισμού 2013, επιβεβαιώνεται ότι θα είναι μια μεγάλη πολιτική δυσκολία και η σύμπτωση του χρονοδιαγράμματος ε, οδηγεί στο ότι στην πράξη θα διαπραγματευτούμε το ύψος των πληρωμών του των πιστώσεων πληρωμών του 2013 ταυτόχρονα με το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Εμείς θέλαμε να τα αποφύγουμε. Θα θυμάστε ότι πολλές φορές είπαμε στις διάφορες διαδοχικές προεδρίες, Πολωνική, Δανέζικη, Κυπριακή και τώρα στην Ιρλανδική, και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι έπρεπε εκ πάση θυσία να προσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μην περιπλακούν οι διαπραγματεύσει αυξάνοντα το πακέτο. Τώρα όμως έτσι έχουν συμπέσει τα χρονοδιαγράμματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε να ε, να μειχθούν οι διαπραγματεύσει, ε, δεδομένου ότι υπάρχει και ένας άμεσος, ε, μια άμεση συσχέτιση, εφόσον όσα δεν πληρωθούν το 2013 θα πρέπει να πληρωθούν το 2014. Και δεδομένου του τι συνέβη πέρυσι, για να υπάρξει δηλαδή αλληλουχία ανάμεσα στο 2012 και στο 2013, είναι προφανές ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, όπως είπε και ο εισηγητής μας. Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών του 2013, το Κοινοβούλιο βασίζεται σε δύο κατηγορίες κειμένων. Πρώτον, τις δηλώσεις που έχουν επισυναυθεί στον προπολογισμό του 2013 και κυρίως την περίφημη δήλωση που είχε επιμείνει να διαβάσει ο ίδιος ο πρόεδρος Σούλτς τη στιγμή της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο δίνοντας ε, προφορικά την, ε, ε, την ερμηνεία που έδινε το Κοινοβούλιο σε αυτή τη δήλωση όσον αφορά τις υποαναστολή πληρωμές suspended payments και τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί πως αυτές οι υποαναστολή πληρωμές θα πρέπει πλήρως να χρηματοδοτηθούν από φρέσκα χρήματα, fresh money. Δεύτερη κατηγορία κειμένου επί το οποίο βασίζεται το Κοινοβούλιο είναι το ψήφισμα της 13ης Μαρτίου στο οποίο είπαμε ξεκάθαρα ότι οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές ε, πλαίσιο δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν να έχουμε ένα σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα μας προτείνει τη ρύθμιση του προβλήματος όλων των απλήρωτων λογαριασμών του 2012 και δεύτερον, στο ψήφισμα αυτό είπαμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές πλαίσιο χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε όλα τα προβλήματα πληρωμών του 2013. Και όταν λέμε να τα ρυθμίσουμε, σημαίνει να τα ρυθμίσουμε χωρίς καμιά εφεύρεση του τύπου υποαναστολή πληρωμέ, αλλά τηρώντα τον δημοσιονομικό κανονισμό, ε, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι λογαριασμοί που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξοφληθούν μέσα σε προθεσμίες που σύμφωνα με τον τρόπο διαχείρισης ή τη φύση της οφειλής συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε έξι μήνες και ε, έξι εβδομάδες και δύο μήνες. Δηλαδή, όλες οι, όλοι οι λογαριασμοί θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή πλέον υποαναστολή πληρωμές, ακόμα και αν τις ονομάσουμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν μέσω αυτού του ψηφίσματος που υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, τρία τέταρτα των ψηφισάντων και αυτό το υπενθυμίσαμε επανειλημμένως σε διμερείς επαφές στο πλαίσιο επαφών με τρεις ή τέσσερις συμμετέχοντες, ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Σούλτς. Η Κομισιόν λοιπόν εργάζεται επί ενός σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού του 2013 με την ιδέα να ρυθμίσει μια ή να ρυθμίσει το μεγαλύτερο τμήμα με ένα σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού το οποίο θα υποβληθεί γρήγορα την Άνοιξη. Είμαστε στις αρχές της Άνοιξης. Και ο πρόεδρος Μπαρόζο χρησιμοποίησε μάλιστα την εικόνα του Big Bang. Μπαίνουμε δηλαδή σε ένα σύμπαν υπό διαστολή διαστολή τώρα δημοσιονομική ή ρητορική θα είναι. Πάντως, η Κομισιόν εργάζεται από αυτού και ο Επίτροπος δεν θέλησε να μας δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία το σύνολο των Επιτρόπων θα εγκρίνει το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού. Το καταλαβαίνω και ο καθένας θα καταλαβαίνει ότι Δεδομένες τις συγκυρίες και του προβλήματος που τίθεται όσον αφορά την απόφαση για την βοήθεια προς τη δημοκρατία της Κύπρου, η Κομισιόν θα προτιμήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για το ειδικό προπολογισμό αλλά θα είναι τώρα κοντά η ημερομηνία αυτή και σε σχέση με βάση μάλλον το περιεχόμενο της πρότασης θα αποφασίσουμε εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις επί του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του διορθωτικού προϋπολογισμού. Τέλο, όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού 2014, εδώ έχουμε μπροστά μας δύο προβλήματα, όπως πολύ καλά το εξήγησε η Άννη Γένσεν. Το ένα είναι θέμα αναφορά και το άλλο είναι το θέμα χρονοδιαγράμματος. Το πρόγραμμα αναφορά είναι το πρώτο ζήτημα που θέτει και που προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί πλέον να βασιστεί στις ε, προτάσεις του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 για να επεξεργαστεί τον προπολογισμό του 2014, γιατί εντωμεταξύ υπήρξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8 Φεβρουαρίου. Όμως η Κομισιόν δεν μπορεί να πάρει ως ε, αναφορά τα νούμερα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει θέση επί της ουσίας, αλλά έχει υιοθετήσει ψήφισμα όπου λέει ότι απορρίπτει αυτά τα νούμερα. Ή μπασπιπτούσε ότι απορρίπτει τα πορίσματα που περιλαμβάνουν αυτά τα νούμερα. Είναι ευθύνη της Κομισιόν λοιπόν να βρει με βάση όλα αυτά την αναφορά που θεωρεί ότι θα αντιστοιχεί Στι ανάγκε και στι δυνατότητε. Αυτή είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο εισηγητή είπε ότι το Κοινοβούλιο όσον το αφορά θα ήθελε φυσικά η αναφορά να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στην αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά το επαναλαμβάνω είναι ευθύνη της Κομισιόν. Δεύτερο, δεύτερη κατηγορία προβλημάτων είναι το χρονοδιάγραμμα. Αρχικά η Κομισιόν είχε προβλέψει σύμφωνα με το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα να εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού προς τα τέλη του Απριλίου και ήμασταν ε, σε φιλική συζήτηση για να δούμε αν θα είναι η παραμονή της Πρωτομαγιάς ή η επομένη ή η ίδια η Πρωτομαγιά αλλά από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση χρονική. Προσανατολιζόμαστε τα τέλη του Μαΐου. Τότε θα υιοθετήσει το σχέδιο της Κομισιόν. Θύμισα στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι που συμφώνησε μαζί μου ότι θα θέλαμε, όπως κάθε χρόνο, ο Επίτροπος Αρμόδιος επί του προϋπολογισμού να έρθει και να, να δημοσία να παρουσιάσει το σχέδιο προϋπολογισμού ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών πριν το σχολιάσει στον τύπο και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε, δεν έχουμε ακόμα πλήρη συμφωνία για όλες τις ημερομηνίε, αλλά για τη συνέχεια της διαδικασίας Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε θεσμικό όργανο θα έχει τον απαραίτητο χρόνο και κυρίω το Κοινοβούλιο θα έχει τον απαραίτητο χρόνο μετά από την ψηφοφορία σε επίπεδο του Συμβουλίου κατά διάρκεια των θερινών μηνών έτσι ώστε η Επιτροπή μας και οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές να έχουν επαρκή χρόνο για να καταθέσουν τροπολογίες, εμείς να έχουμε αρκετό χρόνο για να εξετάσουμε τις τροπολογίες τους και να φτιάξουμε τις δικές μας τροπολογίες τη Επιτροπή Προπολογισμού και οι πολιτικές ομάδες να έχουν στη συνέχεια αρκετό χρόνο ώστε να εκτιμήσουμε, εκτιμήσει την εργασία μας και να λάβει θέση και να διευκρινίσει τη θέση του πάνω στις δικές μας τροπολογίες. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα και εμείς θα τα ξεκαθαρίσουμε κάπως περισσότερο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας έχει ε, παρουσιάσει το διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 1 του 2013. Αυτά. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε εδώ σήμερα τον Γενικό Διευθυντή επί του προπολογισμού της Κομισιόν. Θέλετε κάτι να πείτε, να διορθώσετε. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη σιωπηρή αλλά προσεκτική, προσιλωμένη παρουσία του Γενικού Διευθυντή. Continuons. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε στο πλαίσιο της παρουσίασης του προϋπολογισμού 2014 με το έγγραφο εργασίας που αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχει διανεμηθεί. Αν θέλεις να το σχολιάσεις για το, τα πιλωτικά προγράμματα και ο Τζοβάνι και οι δυο, η Το έγγραφο εργασίας μας δίνει έναν κατάλογο των πιλωτικών προγραμμάτων. Μας δίνει μια επισκόπηση μάλλον των όσων ήδη αποφασίστηκαν και έχουμε μια έκθεση της Κομισιόν που εξετάζει τα πιλωτικά προγράμματα που εγκρίναμε για το 2013 όπου η Κομισιόν περιγράφει το πώς θεωρεί ότι θα λειτουργήσουν και ο Τζοβάνι θα μιλήσει γι' αυτό. Εγώ απλά θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τη διαδικασία, έχουμε μια διαδικασία για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ε, δράσεις. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια αρχική, μια προκαταρτική ε, ε, πρόσκληση ε, για υποβολή αιτήσεων, ώστε η Κομισιόν να έχει την ε, δυνατότητα να εξετάσει ε, τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, ώστε να μην, να έχουμε προτάσεις που να καλύπτονται από τις υπάρχουσες νομικές βάσεις. Οι προτάσεις μη σκόπιμες. Τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις όπως ε, θα θυμούνται οι ευρωβουλευτές, είναι προγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει νομική βάση. Το πιλωτικό πρόγραμμα στόχο έχει να δοκιμάσει νέες ιδέες, οι προπαρασκευαστικές δράσεις επικεντρώνονται περισσότερο στην προετοιμασία της νομοθεσίας ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν οι γραμμές του προϋπολογισμού προτού να υπάρχει νομική βάση και έχουμε διάφορα παραδείγματα όπου το Κοινοβούλιο δημιούργησε νέες ιδέες, οι οποίες τώρα αποτελούν μέρος των ευρωπαϊκών πολιτικών, όπως είναι το Ταμείο Προσφύγων και άλλα πράγματα. Έχουμε αρκετά πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις και αυτό μας δείχνει ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για προγράμματα που οδηγούν σε νέες πολιτικές, σε νέα νομοθεσία ή που να προδικάζουν τη νέα νομοθεσία. Πότε πότε. Βλέπουμε οι Ευρωβουλευτές ή ακόμα και η Κομισιόν να θέλει να αναλυφθούν δράσεις σε περιοχές όπου δεν υπάρχει, σε τομεί όπου δεν υπάρχει η νομική βάση και που μπορεί να χρειάζεται χρηματοδότηση για ένα-δύο χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν κάποια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως αργότερα να μπορούν να κάνουν μόνοι τους σε τομείς όμως που να μην καλύπτουν από τους πόρους που ήδη διατίθενται. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τις πολιτικές μας με ιδέες, να δοκιμάσουμε νέες ιδέες με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει ε, ένα όριο 40 εκατομμύριων ευρώ για τα πιλωτικά προγράμματα. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το όριο του χρόνου, διότι δεν έχουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ακόμα. Μπορεί να παραμείνει το ίδιο το ποσό αυτό, μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ ή μπορεί να μειωθεί. Δεν νομίζω ότι θα δεχόμαστε να γίνει μείωση, αλλά για τα πιλωτικά προγράμματα 40 εκατομμύρια, τις προπασκευαστικέ δράσεις έχουμε 100 εκατομμύρια συνολικά και μόνο τα 50 εκατομμύρια μπορεί να καλύψουν νέες ιδέες. Επισκέφτομαι τις εξειδικευμένες ε, επιτροπές αυτή τη στιγμή και τους ε, ενημερώνω να ε, έχουν κατά νου την προθεσμία τον Μάιο. Σε κάποιους τομείς Μπορεί να έχουν ε, διάφορες ιδέες. Ε, η Επιτροπή Μεταφορών έχει χρησιμοποιήσει τα πιλωτικά προγράμματα για να χρηματοδοτήσει τουρισμό, διότι ο τουρισμός συμπεριλαμβάνεται ε, στην συνθήκη, δεν υπάρχει όμως ειδική γραμμή του προϋπολογισμού. Και αυτό μας δείχνει πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σχετικά μικρά ταμεία για να ε, υποστηρίξουν πολιτικές ε, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ε, ειδικέ γραμμές του προϋπολογισμού. Οι παρατηρήσεις της Κομισιόν είναι φυσικά σημαντικές και θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας κατά τη συζήτηση για το αν θα πρέπει να παραταθεί ή να, προωθηθεί, να ένα πρόγραμμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε συζήτηση με τις ειδικέ επιτροπές σχετικά με τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και το πώς λειτουργούν, διότι μερικές φορές απαιτείται διάλογος ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο στόχος και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Όταν, συμμετείχα, όταν παραβρέθηκα στην ε, Επιτροπή Γεωργίας, αναφέρθηκε ε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τις γεωργικές τιμές και το τι γίνεται στην ε, αλυσίδα από τον αγρότη μέχρι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις σχετικά με το τι ακριβώς αναζητούμε και γι' αυτό μπορεί να διαφέρει η αξιολόγηση της Κομισιόν από την αξιολόγηση του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο ω Επιτροπή του Υπεροπολογισμού να βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους ανθρώπους που ζήτησαν τα πιλωτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίσουμε να γίνει σωστά η εφαρμογή. Να ακούμε λοιπόν την Επιτροπή, να, ακούμε όμως και τους συναδέλφους μας. Νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο και σωστό. για τις επιτροπές και τους ευρωβουλευτές ε, λέμε ότι η προθεσμία είναι τέλη Μαΐου και τον ε, Ιούνιο θα γίνει η αξιολόγηση. Και αφού ακούσουμε τις απόψεις της Κομισιόν θα μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Ευχαριστώ πολύ, Άννο Τζοβάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για τον προπολογισμό 2013 οι συνάδελφοι υπέβαλαν 142 προτάσεις πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων και καταφέραμε, μάλλον αποφασίσαμε, να εισάγουμε 58 από τις οποίες 27 είναι πιλωτικά προγράμματα και 31 προπαρασκευαστικές δράσεις στο ε, δημοσιονομικό σχέδιο του προπολογισμού. Η Άννα ε, μας ανέφερε ποιο ήταν το ποσό που προβλεπόταν στη Διαθεσμική Συμφωνία και στην πράξη εμείς ε, χρησιμοποιήσαμε ένα επίπεδο πόρων σαφώς χαμηλότερο σύμφωνα με αυτό που ήταν ε, η συμφωνία, η συνεννόηση να μειώσουμε όσο γίνεται τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές μέσα στον προπολογισμό του 2013. Για τα πιλωτικά προγράμματα σε σχέση με ένα ανώτατο όριο 40 εκατομμυρίων χρησιμοποίησαμε μόνο 22,2 και για τις ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις και 31 για τις πληρωμές. Και όσον αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, για τις 31 προπαρασκευαστικές δράσεις που βάλαμε στο πακέτο, χρησιμοποιήσαμε 49,9 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις και 61 στις πληρωμές. Για το πλαίσιο της έκθεσης που υποβάλλουμε σήμερα με τη συνάδελφο Αν, υπάρχουν κάποιες βέβαια λεπτομέρειες περισσότερες όσον αφορά την κατανομή ανά τίτλο του προϋπολογισμού Κάτι που θέλω να θυμίσω και είναι σημαντικό νομίζω να το κάνω σήμερα. Να σας θυμίσω λίγο τη διαδικασία. Η Κομισιόν έχει υποβάλει την πρώτη ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων στις 28 Φεβρουαρίου του 2013 και αυτό το έχουμε εντάξει στον προγραμματισμό και αυτό προφανώς μας ε, δίνει ένα μικρό περιθώριο όσον αφορά την πρόοδο των προγραμμάτων που έχουν ε, ε, συμπεριληφθεί στην προηγούμενη χρήση και στον προϋπολογισμό του 2013. Είναι σαφές ότι θα το συζητήσουμε και ότι θα έχουμε επαφές με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ώστε ο καθένας να δει πού βρίσκεται η διαδικασία, η πορεία που προβλεπόταν για τα προγράμματα που έχει υποβάλει. Επόμενο βήμα θα είναι να παρουσιαστεί η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση για τα πιλωτικά προγράμματα που προβλεπόταν για τον Απρίλιο του 2013 και εδώ θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω την Κομισιόν εφόσον προβλεπόταν από κοινού με την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού αν και αυτό θα διολυστήσει όπως προβλέπεται και η προϋπολο... όπως και ο προϋπολογισμός ή αν θα πρέπει όντως να το περιμένουμε τον Απρίλιο του 2013. Τώρα, σε σχέση με τη διαδικασία, νομίζω πως είναι προφανής η ανάγκη όσοι έχουν υποβάλει προγράμματα να κάνουν ένα διάλογο με την Κομισιόν ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία εφαρμογής και για να στηρίξουν την πρόοδο των πιλωτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών ε, δράσεων. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε και εν ώψη της ε, παρουσίασης νέων πιλωτικών προγραμμάτων και προπαρασκευαστικών δράσεων ότι έχουμε πολλά πιλωτικά προγράμματα που με το 2013 βρίσκονται στο δεύτερο έτος εφαρμογής τους και άρα θα χρειαστεί ή να μετατραπούν σε προπαρασκευαστικές δράσεις στον επόμενο προπολογισμό είτε απαιτείται για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι δραστηριότητές τους να μετατραπούν μέσω πρωτοβουλία πρωτοβουλίας της Επιτροπής σε μια νέα ε, νομική βάση. Επίσης έχουμε διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις που βρίσκονται στο τρίτο έτος εφαρμογής και που άρα ακόμα δεν μπορούν να παραταθούν στην σχετική δραστηριότητα και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να υπάρξει δυνατότητα εφαρμογής μιας νέας νομικής βάσης αν χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι ακόμα όσον αφορά τις πιλωτικές, τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που είναι υπό εξέλιξη. Ευχαριστώ. Τζοβάνι Αίντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ περίεργο να βλέπουμε πόσο αυτά τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσει που είναι ένα μέσο που έχει πολύ μικρό προπολογισμό αλλά δημιουργεί πολύ ενδιαφέρον νομίζω με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε ε, άλλους βουλευτές από άλλες επιτροπές να καταλάβουν καλύτερα τον προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή που λύγει η θητεία θα έπρεπε να κάνουμε μια πιο αναλυτική αποτίμηση όχι μόνο αυτών που διεξάγονται αυτή τη στιγμή αλλά και όλων όσα έλαβαν χώρα για αυτές τις ενέργειες ε, ποια πήγαν καλά, ποια όχι πόσα ε, προκάλεσαν ε, νομοθετήματα της Ένωσης εάν οι στόχοι τους ήταν διαφορετικοί ή ευρύτεροι από ό,τι περιμέναμε. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια μελέτη που θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για να δούμε πώς, πήγε, πώς πήγαν αυτές οι ενέργειες σε αυτή τη θητεία και ίσως την επόμενη να έχουμε έτσι έναν απολογισμό του τι έχει συμβεί, τι προβλήματα υπήρξαν και τι λύσεις. Διότι τα προγράμματα αυτά, τα πιλωτικά και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες είναι στην ουσία δοκιμή των προσεχών ευρωπαϊκών πολιτικών και άρα πρέπει οπωσδήποτε να αποτιμήσουμε τι έγινε. Ευχαριστώ. Λαμασού. Ευχαριστώ, Ειντερ. Θα ήθελα και εγώ να πω, όπως είπε και η Ειντερ, ότι αυτή η διαδικασία πιλωτικά και προπαρασκευαστικές ενέργειες θα έχει μεγάλο αντίκτυπο το 2014 που είναι εκλογικό έτος και για το παρελθόν δηλαδή και για το μέλλον δηλαδή για το παρελθόν όπως είπε η Ειντερ, θα είναι μάλλον ενδιαφέρον στο τέλος της θητείας να κάνουν απολογισμό του τι μας επέτρεψε αυτή η διαδικασία που όπως θα θυμάστε δημιουργήθηκε ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει δυνατότητα να εκκινήσει μερικές πολιτικές πρωτοβουλίες σε τομείς που δεν έχουμε ακόμη νομική βάση για να προωθήσουμε τις ε, νομικές πρωτοβουλίες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σωστά λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε εάν το Κοινοβούλιο μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή τη διαδικασία για να ευρύνει την ε, δραστηριότητα της Ένωσης, να εντείνει και να επιταχύνει τη δράση μας σε τομείς που είναι αρμοδιότητα της Ένωσης, αλλά, αλλά όπου η Επιτροπή δεν είχε ακόμα να λάβει πρωτοβουλίες. Ε, νομίζω ότι οι συγητές μας άκουσαν αυτή την πρόταση και θα τη λάβουν υπόψη. Με κάποια μορφή. Το 2014 ε, όμως είναι και η απαρχή μιας νέας περίοδου. Διότι, διότι έχει ε, τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας που χορηγεί νέες αρμοδιότητες ή διευρύνει υπάρχουσες για την Ένωση. Υπάρχουν τομείς λοιπόν όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες. Θα μπορούσαμε λοιπόν, για πολιτικούς λόγους, διότι κάποια πολιτική ομάδα ενδιαφέρεται για την α ή β πολιτική ή γιατί το κοινοβούλιο συνολικά θέλει να αναπτύξει περαιτέρω την αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα της Ένωσης, μπορεί λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ε, διαδικασία για να αξιοποιήσουμε καλύτερα το νομοθετικό δυναμικό των συνθήκων. Για παράδειγμα, η Άννα ανέφερε τον τομέα του τουρισμού, που τώρα όμως είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Βεβαίως, για πολλές χώρες είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα και σε περιοχές της Ισπανίας, για παράδειγμα, στη χώρα των Βάσκων. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, για παράδειγμα, το διάστημα. Βεβαίω, πιλωτικό πρόγραμμα για το διάστημα, ωραία ιδέα. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία θεμάτων. Μια άλλη θα έλεγα. Που ενδιαφέρει ίσως περισσότερο το Συμβούλιο. Διότι αυτή η διαδικασία πιλωτικών προγραμμάτων βεβαίως μπορεί να αξιοποιηθεί και από τα δύο σκέλη τη αρχή προπολογισμού μέχρι στιγμή την έχει αξιοποιήσει. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει και το Συμβούλιο. Για παράδειγμα, των δώρων. Gifts, λίγο άθλιων, που αναφέρονται στα πορίσματα του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου στα πλαίσια των πολιτών προοπτικών εκεί, στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποιες επιταγές κάποιου είδους που θα μπορούσαν να ζωθούν σε κάποιες χώρες χωρίς καμία συνθήκη, καμία προϋπόθεση. Οι χώρες παραλήπτες βεβαίως ε, χαίρονται ιδιαίτερως. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, θα το έβρισκαν καλό αν έλαβαν ο καθένας τέτοιο, τέτοια επιταγή, τέτοιο τσεκ. Αλλά επειδή είμαστε χώρος δικαίου, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλήρε αρμοδιότητε για δημοσιονομικά θέματα, για τον ετήσιο προπολογισμό, τουλάχιστον όσον αφορά τις δαπάνες. Οπότε, δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε ότι θα δώσουμε ένα ποσό σε μια χώρα, μια περιφέρεια, μια επιχείρηση, ένα άτομο, μια τρίτη χώρα, χωρίς νομική βάση χωρίς αιτιολόγηση. Να τους δώσουμε κάποιο ποσό γιατί η χώρα αυτή και τα λοιπά έχει κάποιες δυσχέρειες ή ε, θέλει να αναλάβει ένα σημαντικό πρόγραμμα, μια σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη της Ένωσης, των αξιών της Ένωσης τα Πρέ, πρέπει να αιτιολογήσουμε. Αν αιτιολογήσουμε είναι ρουσφέτη είναι το αθλιότερο επίπεδο της πολιτικής ζωής. Έχω πολιτικούς φίλους, τους χαρτζηλικώνω. Έτσι λειτουργήσε το Συμβούλιο, μου φαίνεται, σε έναν βαθμό τουλάχιστον. Και γι' αυτό, εσκεμένα, χρησιμοποιώ τον όρο ότι είναι άθλια αυτά τα πράγματα. Και εμείς ως Κοινοβούλιο πρέπει να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τέτοιου τύπου ενέργειες για να επιτευχθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο για το δημοσιονομικό πλαίσιο ήταν ε, κατανοητό πριν τη Λισαβόνα, ήταν παράδοση, γινόταν, το καταλαβαίνουμε. Τώρα πλέον δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν μάλιστα, κυρίως, ενώ επίκυνται ευρωεκλογέ, όπου θα πρέπει να κάνουμε απολογισμό, όπου ο καθένας μας μπορεί να αντιμετωπίσει ερωτήσεις για το πώς πήγαν οι διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί δεχθήκατε να δοθούν 200-300 εκατομμύρια στην Α χώρα και όχι στη Β. Θα πρέπει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε. Σε πολλές γλώσσες αυτό λέγεται κράτος δικαίου. Είναι το αντίθετο της αυθαιρεσίας. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αιτιολογούμε τις ενέργειές μας. Το πρόβλημα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε στη διαπραγμάτευση. Και το αναφέρω όχι γιατί θέλω να περιπλέξω τη διαπραγμάτευση. Όχι καθόλου. Δεν θέλω να ενοχλήσω το Συμβούλιο. Όχι. Αλλά γιατί πρέπει όλοι από κοινού να καταλήξουμε σε λύση που να μπορέσουμε να αιτιολογήσουμε έναντι των πολιτών και εκλογέων. Τα υπενθυμίζω και προς τους εισηγητές μας, διότι και ιδίω τον εισηγητή του πολιετού πλαισίου, γιατί θα μπορούσε να αξιοποιήσει ε, τα στοιχεία αυτά για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Θα ήθελα να σχολιάσουν οι Όχι, όχι. Όχι, ούτε η Άν, ούτε ο Τζοβάνι. Οπότε ευχαριστώ. Ακούσατε λοιπόν ποιες είναι οι προθεσμίες από τους εισηγητές μας και ο Τζοβάνι έθεσε ερωτήματα στην Κομισιόν και θα λάβει απάντηση. Οπότε, να δώσω το λόγο στην Αν Γένσεν για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης για την ε, υλοποίηση ενισχυμένης συνεργασίας για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να επαναλάβω το λόγο που έχουμε την πρόταση αυτή. Έχουμε πρόταση από την Κομισιόν για φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και η Επιτροπή μας αξιολόγησε την ε, πρόταση και συμφώνησε ότι πληρεί τα κριτήρια ε, για, ίδιου, για τους ίδιους πόρους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιοι. Και αυτό συμπεριλήφθηκε στην ε, γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ που ε, γνωμοδότησε και υπήρχε και ε, πλειοψηφία εντός του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν είχε πλειοψηφία και χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο μάλιστα και γι' αυτό βρισκόμαστε στη θέση 11 χώρες να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ε, για μια ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά τον ε, φόρο επί των χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Και η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση για ενισχυμένη συνεργασία πάνω στο θέμα αυτό. για 11 χώρες. Ουσιαστικά, Πρόκειται για την ίδια πρόταση με πριν, αλλά με μια μικρή τροποποίηση όσον αφορά όχι μόνο ε, το, τον μόνιμο κάτοικο, αλλά και την ε, ε, αλλά και, ε, ε, και το είδο, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να επηρεάσει και τα σταξιδοτικά ταμεία και ανθρώπου που ζουν εκτό των 11 αυτών χωρών. Το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι αν πιστεύουμε ακόμα ότι η πρόταση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, πληρεί τις προϋποθέσεις για τους ίδιους πόρους. Και εγώ αυτό προτείνω. Εάν τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία αποφασίσουν ότι ε, εν μέρη ή ολικώς ε, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ε, έσοδα από τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για να μειώσουν τις εθνικές τους συνεισφορές, μπορούν να το κάνουν. Όσον αφορά το πώς θα γίνει αυτό τελικά, στις σελίδες 19 και 20 της έκθεσης, Το θέμα είναι αν κάθε χώρα θα πρέπει να αφαιρεί το δικό της μερίδιο από το ποσό ή αν θα πρέπει να συγκεντρώνονται τα έσοδα και κατόπιν να μειώνεται ε, η συνεισφορά του ακαθαρίστου εθνικού εισοδήματος ε, του εν λόγω κράτους μέλους. Υπάρχουν δηλαδή δύο διαφορετικές αρχές, είτε να συγκεντρώνουμε τα έσοδα ή να αφαιρούμε από το μερίδιο της κάθε χώρας. Ε, δεν έχω αποφασίσει ακόμα ποια μέθοδος θα είναι πιο σκόπιμη. Αυτό είναι το βασικό θέμα της γνωμοδότησης που υποβάλλουμε προς την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι ε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, διότι ουσιαστικά δεν αλλάζει το σύστημα που ήταν η πρόθεση με την αρχική πρόταση. Και πάλι δηλαδή θα μιλάμε για εθνικές συνεισφορές και τη μείωσή τους. Αλλά αυτά θα υποβάλω στην Επιτροπή και θέλω να ακούσω τις, ε, τη γνώμη των ε, Ευρωβουλευτών της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζαν ο πρόεδρο εκ παραδρομή. Ε, Άννα, ευχαριστώ. Αλλά επειδή και ο Ζαν είναι συνηγητή, θα πρότεινα να πάρει πρώτα το λόγο ο Ζαν και μετά ούτε και οι άλλοι ομιλητέ. Νομίζω ότι. En grande ligne, euh, la proposition que la... Βλέποντα την πρόταση που είχε κάνει η Κομισιόν για το σύνολο των κρατών μελών και στην γνωμοδότηση της αν συμπεριλαμβάνεται και η γνωμοδότηση που είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά. Πάντως το κεντρικό σημείο είναι αυτό που ανέφερε στο τέλος της ομιλία τη. Για μένα είναι σαφές ότι αν μιλάμε για ίδιους πόρους δεν υπάρχει παρά μόνο μία εναλλακτική. Δηλαδή έχουμε έναν πόρο που είναι ευρωπαϊκός και μειώνουμε κατά μέσο όρο την συμβολή από το εθνικό ε, καθαρίστο προϊόν. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν, ε, δεν στέκει το ίδιο το πνεύμα του ίδιου πόρου. Επ' αυτού πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, πολύ σαφείς, γιατί μάλιστα πιστεύω ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν έχει μεγάλο νόημα αν απλά ο στόχος είναι να μειωθεί η εθνική συνεισφορά με τα όσα αποδίδει ο φόρος σε εθνικό επίπεδο. Γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουμε από το σύστημα, μένουμε στο ίδιο σύστημα που ισχύει και σήμερα. Και από αυτό θα πρέπει η Κομισιόν να είναι σαφής. Γιατί διαφορετικά θα αποκλίνουμε και όλη αυτή η συζήτηση θα έχει νόημα. Ε, Ευχαριστώ, Ζανλίκ. Η Ούτα. Θα Ήθελα να ε, συμφωνήσω κατά κάποιο τρόπο με τον Ζων Λουκ, διότι βλέπω ότι προσπαθείτε να κάνετε με τις ε, τροπολογίες σας. Ε, έχετε συμπεριλάβει αυτά που είχαμε εγκρίνει με την έκθεση Ποδηματά. Και η τροπολογία 2 είναι αντιγραφή από την έκθεση αυτή. Αλλά έχουμε και το ψήφισμά μας ε, της 13ης Μαρτίου, όπου λέμε σαφώς ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα μέρος των εσόδων των φορολογικών εσόδων ε, να θεωρούνται οι ίδιοι πόροι. Και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να τονίσουμε κάπως περισσότερο αυτήν την τροπολογία. Αυτά που είπαμε στο ψήφισμά μας, ε, να τα επαναλάβουμε, να τα τονίσουμε και να πούμε ότι ο στόχος ε, είναι ακριβώς ε, είναι ο στόχος είναι να μειώσουμε τις μεταφορές πληρωμών από τα κράτη-μέλη. Διότι εξαρτώμαστε συνέχεια από, τις, από τη μεταφορά χρημάτων από τα κράτη-μέλη. Ε, και τα κράτη-μέλη μας λένε ότι σας δίνουμε τα χρήματα και κάπως έτσι εξαφανίζεται, ξεχνιέται η νομική υποχρέωση και αυτό το θέμα θα το λύσουμε μόνο εάν έχουμε οι ίδιους πόρους. Δεν μπορούμε τώρα να φορτώσουμε ε, υπερβολικά την έκθεση αυτή, αλλά πέρα από αυτήν θα ε, επιμείνουμε να έχουμε ίδιους πόρους ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ε, μεταφορά των, ε, τις συνεισφορές των κρατών μελών, αυτό το μερίδιο δηλαδή του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Ίσως ε, θα μπορούσαμε μαζί να κοιτάξουμε λίγο την τροπολογία 2, να τονίσουμε περισσότερο τη διατύπωση, ώστε να ακολουθεί περισσότερο την κατεύθυνση του ψηφίσματός μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ισαβέλ Τυρό. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ στην υπογράφω προφανώ αυτή την έκθεση. Βρισκόμαστε σε ένα είδος ε, ε, πορείας του έχτερνα όσον αφορά αυτό το θέμα. Προχωράμε σιγά σιγά Επιτέλους ε, καταφέραμε για τις 11 χώρες και ήθελα να είμαι βέβαιη, ε, ε, Άννα, ότι η μείωση των εθνικής συμβολής δεν θα ισχύσει παρά για όσους συμμετέχουν στην φορολόγηση για τις εν λόγω 11 χώρες, όχι να υποφεληθούν και οι υπόλοιποι. Επίσης να δούμε το κίνδυνο ε, τελικά αυτό δεν είναι ίδιο πόρο, αλλά απλά συμβάλλει στο να μειωθούν οι εθνικέ συνεισφορέ. Είμαστε σε μια κλίδα 1 τρίτο προ 2 τρίτα, ε, που θα μα επιτρέψει να έχουμε γύρω στα 15 δις ευρώ. Ε, δεν είναι αμεληταίο με 11 μόνο χώρε. Αξίζει τον κόπο, πιστεύω, αν και πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα για τους άλλους ίδιου πόρους και για το γεγονός ότι δεν είναι μόνο αντιστάθμιση μα στι εθνικέ συνεισφορέ. Προχωράμε σιγά και αργά, αλλά πάντως προχωράμε. Πιστεύω ότι είναι καλό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ιζαμπέλ Χουάνο Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ζαν Λίκ Ιάν Γένσεν. Τι έχουμε μπροστά μας. Έναν εναρμονισμένο εθνικό φόρο για 11 χώρες και που θα πρέπει να έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με όσα συμβάλλουν αυτές οι χώρες από το ΑΕΠ τους. Ουδέτερο, μηδενικό δηλαδή. Με αυτό τον φόρο λοιπόν δεν δημιουργούμε έναν συγκεκριμένο ίδιο πόρο. Τα εθνικά Υπουργεία Οικονομικών λαμβάνουν έναν εθνικό πόρο και τον ε, μεταφέρουν στην Ένωση, μειώνοντας έτσι το ΑΕΠ, το τμήμα του ΑΕΠ που μεταφέρουν. Άρα για τα κράτη-μέλη είναι ουδέτερο, μηδενικό το αποτέλεσμα. Τι δημιουργούμε λοιπόν. Δημιουργούμε ένα είδος ειδικού ΦΠΑ ενός ε, ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Είναι κάτι ανάλογο αυτού που κάνουμε όταν μεταφέρουμε ένα τμήμα του ΦΠΑ στην Ένωση. Αυτή την οδό πρέπει να βαδίσουμε, αλλά να μην ε, απατώμεθα. Τα κράτη-μέλη είναι σε θέση ενδεχομένω να τροποποιήσουν το τι συμβάλλουν στον προπολογισμό ανάλογα με το τι είδου πόρου μεταφέρουν στον προπολογισμό της Ένωσης. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ναι, όντως πρέπει να συνδυάσουμε τις λογικές ε, ανησυχίε των κρατών μελών, ιδίως ε, στην περίοδο αυτή τη τόσο μεγάλης ε, δημοσιονομική πίεση και του αιτήματό μας για επιστροφή σε ίδιου πόρους. Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα είναι σημαντικός και από άποψη αρχή, όπως ε, υπενθύμησαν διάφοροι από εσά. Ως πρώτο παράδειγμα αυτού που θα μπορούσε ενδεχομένως να επαναληφθεί και που θα έπρεπε αργά ή γρήγορα να γίνει και για άλλους πόρους. Διότι είναι σαφές ότι η χρηματοδότηση του ενωσιακού προϋπολογισμού σε μεγάλο βαθμό με ίδιους πόρους, για παράδειγμα της τάξης του 60% όπως προτείνει η Κομισιόν και όπως συμφωνούμε, θα επιτευχθεί μέσω πλέον του ενός φόρων. Αν θέλετε να πείτε τίποτα. Έχει δίκιο η Γιούτα, λέει η Άννε. Ήταν στο ψήφισμα. Οπότε μας δεσμεύει. Είναι απόφαση της Ολομέλειας. Βεβαίως θα το συμπεριλάβουμε στην έκθεση, να δούμε βέβαια τη διατύπωση. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι θα περπατήσει. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε και άλλες καινούργιες ιδέες ιδίων πόρων, αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας στον τομέα των ίδιων πόρων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Θα εξετάσω τις τροπολογίες που θα υποβληθούν και θα προχωρήσουμε. Πρόεδρος. Ωραία. Ευχαριστώ κυρία Συγκήτρια. Ακούσατε τις ε, προθεσμίες για την υποβολή τροπολογιών. Οπότε τώρα θα περάσουμε στο σημείο 9. Προετοιμασία προπολογισμού 14 πάντα. Αλλά τώρα είναι το προσχέδιο για τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Η Μόνικα Χολμάια. Έγινε μια ε, συνδιαλλαγή έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Χολμάιερ. Συνάδελφοι, ήταν κάπως περίπλοκη η διαπραγμάτευση. Μέχρι τελευταία στιγμή χρειάστηκαν συζητήσεις. Βεβαίως, διαπραγματευτήκαμε με 27 κράτη-μέλη, αλλά το βασικό είναι να έχουμε συμφωνήσει εμείς για το δικό μας προϋπολογισμό στην πράξη εδώ και δύο χρόνια έχει παγώσει ο προπολογισμό. Εν τω μεταξύ όμως είμαστε νόπιον ε, μιας ε, χρονιά, όπου λόγω της θητείας προκύπτουν ιδιαίτερα, ιδιαίτερες δαπάνες. Θα γίνουν εκλογές, κάποιοι συνάδελφοι θα φύγουν, κάποιοι νέοι συνάδελφοι θα έλθουν, γύρω στο 50% θα ανανεωθεί το κοινοβούλιο, άρα υπάρχει κάποιο μεταβατικό κόστος. Και κατόπιν Κόστος για τις συντάξεις. Η διαφορά από τις προηγούμενες περιόδους είναι ότι για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη για τους βουλευτές του. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Στις προηγούμενες ε, εκλογικές χρονιές ήταν εν μέρη τα εθνικά κοινοβούλια που έδωσαν μεταβατικές πληρωμές και κάποιες ε, πληρωμές μισθών και συντάξεων. Τώρα όμως έχουμε καθεστώς των βουλευτών, έχουμε καθεστώς των βοηθών. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει μεγαλώσει πια. Έχει γίνει οικονομικά αυτόνομο. Όμως αυτό σημαίνει επιπλέον οικονομικές σκοτούρες και δαπάνες. Ήδη το πέρασμα από τη μία στην άλλη κοινοβουλευτική θυμία σημαίνει αύξηση 2,2% δαπανών που είναι νομικά δεσμευτικές. Δεν προσετέθη κάτι που θέλουμε να λάβουμε ευχαρίστως. Είναι νομικές υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με, την, με τα ε, κίνηση από το ένα... Ε, από το ένα κοινοβούλιο στο άλλο. Επίσης μετά έχουμε ένα ποσό λόγω της ανόδου των μισθών είναι και αυτές νομικές υποχρεώσεις των συνεργατών μας, των υπαλλήλων μας. Οπότε έχουμε μια αύξηση γύρω στο 3,3% καθαρά νομικών υποχρεώσεων λόγω του τέλους της θητείας. Όλες οι άλλες δαπάνες και προστίθεται και κάτι λόγω της ε, ένταξης της ε, Κροατίας οπότε πρέπει να υπολογίσουμε κόστος για όλο το χρόνο, το 2014 και ε, στην ουσία ο υπόλοιπος προϋπολογισμός μειώνεται. Δηλαδή δεν ακολουθεί καν τον πληθωρισμό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένες περικοπές, ιδιαίτερα σημαντικές. Πρόκειται να γίνουν στον τομέα της μετάφρασης. Αυτό το έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ ημών. Αλλά θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε να μην θίξουμε την αρχή της ε, πολυγλωσσίας αλλά μόνο όπου είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν να υπάρχει μετάφραση κατόπιν αιτήματος. Για παράδειγμα, για τη μετάφραση στην Ολομέλεια. Έκανε, κάναμε ε, για ένα χρόνο ένα τεστ και δεν ζητήθηκε καμία γραπτή μετάφραση των εργασιών της Ολομέλειας. Ούτε μία. Οπότε Επιπλέον, θα επιδιώξουμε και άλλες διαρθρωτικές δυνατότητες εξοικονομήσεων ή αναδιαρθρώσεων. Έχουμε αυτό το καθήκον από την κοινή ομάδα εργασίας και η διοίκηση του Κοινοβουλίου έχει αναλάβει το καθήκον να μας υποβάλει προτάσεις σε 7 διαφορετικούς τομείς. Θα τις αναλύσουμε, θα τις συζητήσουμε, θα δούμε αν θα τις εγκρίνουμε ή όχι και τι συγκεκριμένα θέλουμε. Για του χρόνου τρεις τομείς θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα όπου μπορεί να αλλάξουν τα στοιχεία μέχρι το Σεπτέμβριο. Ξέρετε ε, ότι συζητάτε αυτή τη στιγμή το καταστατικό των υπαλλήλων. Ε, αν θα γίνουν αλλαγές, ε, αν θα γίνουν εντός του 2013 φυσικά θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τον προπολογισμό του 2014. Ένας δεύτερος τομέας είναι οι αλλαγές ε, που και εμείς θέλουμε να κάνουμε σε διάφορες δομές αφού τις συζητήσουμε. Και ο τρίτος τομέας αφορά τη δομή του προϋπολογισμού σε σχέση με τις μεταβατικές δαπάνες και τις συντάξεις. Εδώ γενικά έχει επικρατήσει η άποψη ότι την πέμπτη χρονιά πάντα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση ε, και αν κάνουμε μεγάλη αύξηση λοιπόν την ε, πέμπτη χρονιά και μετά έχουμε μεγάλη μείωση την επόμενη χρονιά δεν είναι η καλύτερη αυτή ε, συνολικά διάρθρωση του, του προϋπολογισμού. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή έχει βγάλει ε, τις συντάξεις από τις δυτικές δαπάνες και τις έχει σε ένα χωριστό σημείο του προϋπολογισμού όπου είναι βεβαίως και η πάλι του Κοινοβουλίου. Όμως δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ειδικό τμήμα του προπολογισμού τα μέλη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό παρακάλεσα την διοίκηση του Κοινοβουλίου με συμφωνία των συναδέλφων στην ομάδα εργασίας ζήτησα όλοι να είμαστε στο ίδιο τμήμα του προπολογισμού. Δεν έχει έννοια να αυξάνεται πολύ το κόστος για κάποιο τμήμα των ε, συντάξεων ε, κάθε πέμπτη χρονιά και μετά να υπάρχει σημαντική μείωση, να έχουμε δηλαδή μεγάλε διακυμάνσει. Επειδή ο προπολογισμό είναι πολύ μικρότερο από τον προπολογισμό τη Επιτροπή, για τα διοικητικά μιλάω πάντα, γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με την Επιτροπή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, που ε, με βοήθησαν για να συντάξουμε το ψήφισμά μας και συμφωνήσαμε ότι συνολικά θα επιδιώξουμε να ε, επιτύχουμε έναν λογικό προπολογισμό. Βέβαια υπήρξαν κάποιες διαφωνίες εάν θα συμπεριλάβουμε και τον πληθωρισμό σε αυτά που θα προτείνουμε εγώ νομίζω ότι πρέπει συνολικά να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν σε όλους τους τομείς πριν αποφασίσουμε από αυτού το φθινόπωρο. Αυτό θα προτιμούσα, αλλά εν πάση περιπτώσει τελικά προέκυψε ένα συμβασμός τον οποίο ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε. Παρ' όλα αυτά θα επιδιώξουμε να βελτιώσουμε τον προϋπολογισμό και νομίζω ότι ήδη ως Επιτροπή Προϋπολογισμών έχουμε επιτύχει ήδη πολλά. Το ψήφισμα έχει πολλές λεπτομέρειες, αλλά γενικά λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε εξοικονομήσεις, θέλουμε να κάνουμε καινοτομίε, αλλά χρειαζόμαστε και έναν επαρκή προϋπολογισμό που να μπορεί να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να λειτουργεί. Γιατί δεν έχει καμία έννοια να ψηφίσουμε έναν επαρκή προπολογισμό και μετά να μα επικρίνουν γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα λόγω έλλειψη πόρων. Και κάτι ακόμη, μία προειδοποίηση. Ο προπολογισμό του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί σε προεκλογικέ εκστρατείε. Γιατί έτσι, στην ουσία, εάν επιδιώξουμε να κατηγορήσουμε ένα τον άλλον κατά την προεκλογική εκστρατεία, τελικά θίγουμε τους πάντες, θίγουμε τη δημοκρατία. Είναι σημαντικό όλοι από κοινού να έχουμε κοινή γραμμή για τον προπολογισμό του, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με βοήθησαν. Ευχαριστώ Μόνικα. Herzog. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες ε, σκέψει από πλευράς των σοσιαλιστών. Πιστεύουμε ότι είναι ε, πολύ σημαντικό η εξοικονόμηση και η καλή χρήση των πόρων να αποτελούν βασικές αρχές. Θέλουμε το 2014, τη χρονιά των εκλογών, ε, να να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες εξοικονομήσεις χωρί όμως ε, να ε, έχει αυτό αρνητικέ συνέπειες στην ποιότητα εργασιών του Κοινοβουλίου και θέλουμε να φροντίσουμε να διατηρήσουμε την πολυγλωσία ώστε ε, ο κόσμο να μπορεί να παρακολουθήσει την προεκλογική συζήτηση. Πρέπει να σεβόμαστε του κανόνε περί προπολογισμού. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτό ισχύει και για όλου του ευρωβουλευτέ και για όλο το προσωπικό. Επίση, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι εργασίε που έχουν ξεκινήσει στην ομάδα εργασίας και χαίρομαι που έχουμε τέτοια μεγάλη πλειοψηφία, διότι αυτή δείχνει ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν ε, ε, καταπολεμούν το ένα το άλλο, αλλά ε, συνεργαζόμαστε για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και χαίρομαι που καταφέραμε να πετύχουμε πρόοδο με το πνεύμα συμβιβασμού. και πιστεύω ότι όλοι έχουν κάνει σημαντικά βήματα εδώ. Και μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό στην Επιτροπή μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αυξήσουμε το κύριο στο Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ. Très bien. Merci beaucoup. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Αν υπάρχουν άλλα σχόλια, σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν η συνέχεια όσον αφορά τις ε, ε, προβλέψεις, ε, ποια είναι η συνέχεια, η ψηφοφορία. Και από εκεί και μετά, φυσικά το Προεδρείο και η Ολομέλεια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εγώ πρέπει να πάω στη διάσκεψη των Προέδρων και θα δώσω την Προεδρία στην Γιούτα Χάουκ και θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες ακριβώς με την έκθεση της Μόνικα. Από τις στατιστικές ε, ψηφοφοριών που ήθελα να κρατάω θα τις χάσω τώρα. Liebe Kolleginnen, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε το σημείο 11 στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση των εργασιών ε, της ομάδας εργασίας. Έκθεση εργασίας της κοινής ομάδας εργασίας ε, για τον προϋπολογισμό. αλλά νομίζω ότι συζητήσαμε όσα είχαμε να συζητήσουμε. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει και το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Και έτσι περνάμε στις ψηφοφορίες. Καταρχήν, μία τεχνική ερώτηση. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, τις έχετε βάλει στις συσκευέ. Ο συντονιστής μου ακόμα όχι. Α, ah, It's Βρίσκεται καθοδόν, ωραία. Ο Σαλοντόρ ήταν κάπως πιο γρήγορος. Μισή ώρα πριν ήταν έτοιμος. Υπάρχει κανείς άλλος που να μην έχει κάρτα ψηφοφορίας. Κανείς, ωραία. Mhm. So, liebe dann fangen wir jetzt an und. Συνάδελφοι, ξεκινάμε με την έκθεση της Μόνικα Χολμάιερ. Πρώτα ψηφίσουμε συμβαστική τροπολογία Α. Εάν την εγκρίνουμε, οι τροπολογίες 3, 4, 5 και 6 της παραγράφου 2 ε, καταπίπτουν. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής πρότασης α. Α. Σας παρακαλώ, το α ψηφίζουμε. Wir, ne, ne? A, also das Alphabet, Christian noch ε, ξεκινάμε από την αρχή του αλφαβήτου. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Φτάνουμε στη συμβαστική τροπολογία Β. Και πρωτού ψηφίσουμε τη συμβαστική αυτή τροπολογία, θέλουμε να ακολουθήσουμε το αίτημα των φιλελευθέρων και να ψηφίσουμε χωριστά. Όχι, όχι. Θα ψηφίσουμε σε δύο μέρη τη συμβαστική τροπολογία Β που όλοι έχετε διαβάσει, την οποία έχουν συζητήσει πάρα πολύ. Στην τελευταία πρόταση λέει με τη φιλοδοξία να ε, παραμείνει η άξιση του προϋπολογισμού πιο κοντά ε, στο ποσοστό του πληθωρισμού. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα μόνο το closer. Θέλουμε να συμπεριληφθεί στη συμβαστική τροπολογία ή όχι. Θέλουμε το closer, πιο κοντά δηλαδή, να συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική τροπολογία. Ποιος λέει ναι. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Τρεις ψήφοι κατά, μία αποχή. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της συμβαστικής τροπολογίας Β υπό τη μορφή που έχει. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Συμβαστική τροπολογία C, γάμα. Α, όχι. Τροπολογία 10, παράγραφος 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 12 έχει αποσυρθεί. Φτάνουμε στη συμβαστική τροπολογία γάμα. Αν εγκριθεί καταπίπτουν οι τροπολογίες 13 και 14 της παραγράφου 7. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7α. Τροπολογία 15 με προφορική τροπολογία, η οποία βρίσκεται όμως στο έγγραφό σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 16 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με μία ψηφοκατά εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 20 και 21 είναι όμοιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Με προφορική τροπολογία φυσικά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά.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 Απορρίπτεται 15 υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 23. Wer dafür? Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ με την προφορική τροπολογία 4 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 καταπίπτει. 29 χωριστή ψηφοφορία, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, μάλλον ε, του κυρίου Χάρτουγκ, το πρώτο μέρος από Notes the High μέχρι Economic Crisis και το δεύτερο μέρος συνεχίζεται από το Calls ε, μέχρι Parliament Budget. Ε, το πρώτο μέρος υπέρ, κατά. Καλά, θα ψηφίσουμε πριν συζητήσουμε αν έχει νόημα. Υπέρ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 36 υπέρ. Μάλλον, ε, ναι, είναι συμβατή υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44. Πω, πω, πολύ δουλεύσαν πάνω σε αυτήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D, δέλτα. Παράγραφος 18 καλύπτει τις ε, τροπολογίες 47, 48 και 49. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής ε, τροπολογίας D, δέλτα, υπέρ. Κατά. αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Συμβαστική τροπολογία ή ε, παράγραφος 19 και καλύπτει τις τροπολογίες 51, 52, 53. Ποιος είναι υπέρ, κατά, συγγνώμη, ανάποδα τα είπε η πρόεδρος, εγκρίνεται. Ούτως ή άλλως εγκρίνεται. Η σειρά δεν ήταν απόλυτα σωστή, αλλά εγκρίνεται. Φτάνουμε στην παράγραφο 20, τροπολογία 54, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στα εκτιμώντας. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται επίσης. Φτάνουμε στην ψηφοφορία πάνω στην τροποποιημένη έκθεση. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε.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 Ε, ο καθένας λοιπόν έχει την άποψή του εξαιρετικά. Wir stimmen ab ähm, über die Zahlung ähm, innerhalb des Globalisierungsfonds. Ψηφίζουμε το θέμα του Ταμείου ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ε, πρόκειται για μια πληρωμή προς την Ιταλία. Υπάρχουν αρκετέ τροπολογίε. Μήπω ε, μπορούμε εν μέρη να ψηφίσουμε, μπορούμε να ψηφίσουμε κάποιες τροπολογίες μαζί, όχι? Δεκατέσσερις ξεχωριστά και τις υπόλοιπες unblock, συμφωνείτε όλοι? Όχι, αν αφαιρέσουμε τη 14, να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες unblock, συμφωνείτε? 2, 3, 4, 5, 6 μαζί μπορούμε να τις ψηφίσουμε. 2, 3, 4 μαζί. Καλά, ψηφι... ξεκινάμε. Τροπολογία 2. Καλά, μέχρι να τα βρούμε θα, τα έχουμε, τελειώσει. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ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 17 dafür, 16 17 υπέρ, 16 κατά. Μικρή διαφορά, αλλά εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ένα εκτιμώντας μία τροπολογία. Ε, ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 1 κατά. Καλά, θα ελέγξουμε.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 Κοιτάξτε, λυπάμαι, αλλά οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ε, μία ψήφο παραπάνω. Α, εντάξει, βγήκε ο Γιώργος, ωραία. Ωραία. Ξέρω. Ξέρω ναι, για την ψηφοφορία. Ισοψηφία 16. Υπέρ και κατά. Απορρίπτεται. Θα έπρεπε να έχουμε αφήσει κι άλλον ένα ψηφίσει. Οπότε, συνολικά η έκθεση, όπως τροποποιήθηκε, Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Και η Μαρία. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ψηφίστε εσείς, γιατί ο Γιώργος είπε όχι. Ο δεν θα ψηφίσει. Ωραία. 30 υπέρ. 2 κατά. Μία αποχή. Τώρα έχουμε μία μεταφορά πιστώσεων για τον προϋπολογισμό. Ο εισηγητής μας είναι ο Τζοβάνι. Αυτό σχετίζεται με τα όσα μόλις ψηφίσαμε για την εφαρμογή την, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε. Βεβαίως, λογικό. Μόλις εγκρίναμε την έκθεση, λέει Πρόεδρος, για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Τώρα πρέπει λοιπόν να θέσουμε και τις πιστώσεις στη διάθεση του Ταμείου αυτού. Ποιο θα ήθελε να συμφωνήσει με τον εισηγητή λοιπόν. Α, και εσείς έτσι δεν είναι. Και εσείς Α, πολύ ωραία. Όλοι εσείς. Θαυμάσια. Ωραία. Είναι κανείς κατά. Ένας. Ωραία. Αποχές. Μία μάλιστα. Εγκρίνεται. Die anderen, die anderen Ε, τα άλλα σημεία για τον προπολογισμό, ο Ντέρεκ. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο μεταφορές που σχετίζονται με την κατάσταση προβλέψεων. Δεν προτείνεται αύξηση του προσωπικού. Δεν υπάρχουν ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις για φέτος. Η πρώτη αφορά το δικαστήριο που θέλει εννέα μόνιμες θέσεις να γίνουν θέσεις έκτακτου προσωπικού. Η δεύτερη αφορά τον ε, διαμεσολαβητή και ναι μεν δεν είναι αυτή τη στιγμή ε, δεν είναι, καλύπτεται αυτή η θέση γιατί παρετήθηκε θέλει έξι ε, έκτακτες θέσεις να γίνουν μόνιμες οπότε καλύπτονται όλα τα κριτήρια που έχουμε θέσει οπότε προτείνω να τις υπερψηφίσουμε Ευχαριστώ. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή μας, αλλά για τα πρακτικά είναι διαφορετική από την ε, κανονική διαδικασία ε, και δεν βλέπω γιατί είναι πήγον και αλλάζουμε ε, το οργανόγραμμα του διαμεσολαβητή χωρίς να υπάρχει διαμεσολαβητής αλλά εν τώρα είναι μικρές αλλαγές θα συμφωνήσω Πρόεδρος, ωραία και τις δύο μεταφορές μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού Συμφωνούμε με τον εισηγητή μας Ποιοι συμφωνούν με τον εισηγητή